Σας ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε την πρώτη έκθεση που είναι η έκθεση του κυρίου Μέντες Δεβίγκο ως προς την απόφαση να μην συγκληθεί συνέλευση για τη μεταρρύθμιση των συνθηκών σε ό,τι αφορά τα μεταβατικά μέτρα για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση το σύνολο της απόφασης, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενο σημείο. Έκθεση Μέντες Δεβίγκο για τα μεταβατικά μέτρα σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τροπολογία 11 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία 11. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 12 καταπίπτει. Τροπολογία 4, ονομαστική ψηφοφορία, Άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Παράγραφος 5. Τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13, νομαστική και πάλι ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίθηκε και αυτή. Τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. έλεγχος, για να είμαστε βέβαιοι. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Ον απορρίπτεται. Τροπολογία 6, ονομαστική. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 8 και 9 καταπίπτουν. Τροπολογία 10. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Ψηφίσουμε το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. The next item on our agenda is the... Επόμενο σημείο της ημέρησης διάταξης είναι πέντε ψηφίσματα για την κατάσταση στην Κυργιζία. We have oral amendment by Ο κύριος Σαλαφράνκα. Προφορική τροπολογία του κυρίου Μπροκ που δυστυχώς κολλείεται σήμερα το πρωί. Πρόκειται για τροπολογία στην παράγραφο 5 που προσθέτει μετά τη μνήα των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, το διαβάζω στα αγγλικά, για να ενισχύσει τη δημοκρατία και την πολιτική απόδοση ευθυνών. Αυτή είναι η προφορική τροπολογία μόνο. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι. Ψηφίζουμε ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη προφορική τροπολογία Το κυρίου Μπαρτολότσι. Προφορική τροπολογία στο σημείο 13. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση, να εξετάσει την ανάγκη ενδεχομένως αποστολής κατεπίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας. Καλώς. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι. Ψηφίζουμε ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το ψήφισμα που έχουν καταθέσει έξι πολιτικές ομάδες για τα ηλεκτρικά οχήματα. Τροπολογία αριθμός 3. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4. Κατά τμήματα ψηφοφορίες. Πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Έχουμε την αναθεωρημένη τροπολογία αριθμός 1. Έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Παράγραφο 6. Έχουμε ακόμα κατά τμήματα ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Εντάξει, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Παράγραφος 7. Έχουμε. Ψηφίζουμε, λέει ο πρόεδρος, υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Τροπολογία 2. Αναθεωρημένη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στο σκεπτικό C, Γ, έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται επίσης. Τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Το επόμενο θέμα είναι ψήφισμα από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων για τις ε, εξαιρέσεις, για τον κανονισμό εξαιρέσεων όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία. Ψη, ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάλι συγχαρητήρια. Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση του κύριου Πέτερλε για την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τη δράση μας κατά του καρκίνου. Ευρωπαϊκή εταιρική σχέση. Αυτό το επόμενο θέμα. Ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επίσης και πάλι συγχαρητήρια στον εισηγητή μας, τον κύριο Πέτερλε. Επόμενο θέμα είναι η ψηφοφορία της έκθεσης της κυρίας Τόγια για κινητοποίηση ενημέρωσης όσον αφορά την ε, διευκόλυνση ενημέρωσης και για την τεχνολογία για την οικονομία χαμηλού άνθρακα. Ξεκινάμε με την παράγραφο 55, κατεβάτα ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας τη ψηφοφορίες. Αποτέλεσμα. Εγκρίνεται. Με 5 ψήφους διαφορά. 304 υπέρ, 299 κατά. Τώρα έχουμε την τροπολογία 61. Α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Παράγραφος 61 υπέρ, κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά και πάλι ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Τόγια λοιπόν. Επόμενο θέμα είναι ψηφοφορία της έκθεσης πρώτη για τη Λευκή Βίβλιο της Επιτροπής «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης». Πριν ψηφίσουμε όμως θέλω να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Πρόντι. Παρακαλώ κύριε Πρόντι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι κλιματικές αλλαγές είναι μια πραγματική απειλή. Μια απειλή που πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Παρά το γεγονός ότι επηρεάζει διαφορετικά ε, τις διάφορες χώρες του κόσμου. Η επιδείνωση πάντως των κλιματικών συστημάτων θα επιδεινώσουν και την οικονομία μας, άρα και τη ζωή των πολιτών. Στο παρελθόν έχουμε ήδη μιλήσει για την κλιματική δικαιοσύνη και την κλιματική διπλωματία ε, τώρα κάτι πρέπει να κάνουμε κιόλα και να μιλάμε με μία φωνή για το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξακολουθήσει να έχει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην δράση μας θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τον ρόλο που παίζουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, τι μπορούν εκείνες να κάνουμε και μαζί τους να συντονιστούμε για να φέρουμε σε πέρας ότι οικονομικές, ή κοινωνικές τενοτομίες πρέπει για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν ε, εταιρικέ σχέσεις ιδιωτικού δημόσιου τομέα ώστε να προχωρήσουν όλες οι πρωτοβουλίες που απαιτούνται κάθε τετραγωνικό μέτρο του, των χωρών μας. Πρέπει ε, να το κοιτάξουμε πάρα πολύ προσεκτικά, να σταματήσει η διάβρωση του εδάφους. Αν χρειάζεται παραπάνω νερό να φροντίσουμε για εδρευτικά έργα με τον τρόπο ο οποίος θα αντιμετωπίσει την διάβρωση του εδάφους και να φροντίσουμε για τις απαιτούμενες προσαρμογές στις νέες καταστάσεις. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που με βοήθησαν στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόντι. Τώρα θα ψηφίσουμε λοιπόν την τροπολογία αριθμό 1 με κατατμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 41. Υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 305 υπέρ, 225 κατά. Πάμε λοιπόν στην παράγραφο 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε και πάλι ηλεκτρονικά. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 3, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 68 τώρα. Υπέρ. Αποχέ. αποχές ας το ανέξουμε παρακαλώ και πάλι ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία voted. Ευχαριστώ ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίθηκε 297 ε, ε, υπέρ 293 κατά πάρα πολύ μικρή διαφορά όντω, είχατε δίκιο η τροπολογία παρθμό 4 ψήφι υπέρ παρακαλώ Against κατά αποχές λεγχός χρειάζεται και πάλι ηλεκτρονικός. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Να ψηφίσατε όλοι. Όχι. Καλά, καλά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τώρα ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Αποτέλεσμα, αυτή τη φορά εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Τώρα, η παράγραφό 73 έχει χωριστεί ψηφοφορία τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εδώ χρειάζεται και πάλι ηλεκτρονικός έλεγχος αρχίζει τώρα η ψηφοφορία Everybody's voted. όλοι πέρας και εγκρίθηκε και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο του σχεδίου όπως τροποποιήθηκε υπέρ από αποχές εγκρίνεται. Και πάλι συγχαρητήρια κύριε Πρόντι. Επόμενο θέμα είναι η ψηφοφορία της εκτίσης του κυρίου Κοτσολίνο για την προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων των κοινοτήτων κατά πολέμηση της απάτης. Θα ψηφίσουμε την τροπολογία υπαριθμών 1 ε, με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ε, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα το σχέδιο ψηφίσματο όπως το και ψηφιπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρτήρι κύριε Κοτσολίν. Επόμενη έκθεση Deutsch. Ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2008. Το ψήφισμα στο σύνολό του ψήφιπε κατά αποχές εγκρίνεται. Και το τελευταίο θέμα σήμερα προς ψήφιση για τις μαζικές θηριωδίες στο Τζος της Νιγηρίας τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο. Νομίζω ότι έχουμε μερικές προσφορικές τροπολογίες. Η πρώτη της κυρίας Κιλ Νίλσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως σας είπα και κατά τη διάρκεια της συζήτησης προτείνω ε, προσθήκη προφορικής τροπολογίας στην παράγραφο περιθμών 6 ως εξής. Καλεί ε, τις αρχές της χώρας να ε, καταργήσουν την πρόσφατη απόφαση ορισμένων κυβερνητών Πολιτειών ε, της Νιγηρίας ε, να εκτελεστούν θανατικές ε, ποινές για να αδειάσουν οι φυλακές από τον υπερπληθυσμό. Αυτό είναι κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλούμε την κυβέρνηση της Νιγηρίας να διατηρήσει το δικαιοστάσιο. Η θανατική ποινή και η εκτέλεσή της είναι αντίθετη με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Νιγηρίας. Any Μάλιστα. Διαφωνεί κανεί. Ψηφίζουμε λοιπόν. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Ο κύριος Κατσμάρεκ τώρα θέλει να κάνει και εκείνο στην παράγραφο 7 τώρα ε, προφορική τροπολογία. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι. Πρόκειται για την ελευθερία της έκφρασης και είναι κάτι που συζητείται και μέσα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και Νιγηρίας στα πλαίσια της συμφωνίας του Κοτονού. Υπάρχουν ενστάσεις; Όχι. Υπέρ. Κατά. αποχές Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος Ψήφι υπέρ. Κατά. αποχές Εγκρίνεται. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η ώρα έχει φτάσει 11.30. Μας μένουν περίπου 25 λεπτά μέχρι ότου προσέλθει ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Μπάιντεν. Προτείνω λοιπόν να ακούσουμε τώρα τις επεξηγήσεις ψήφου μέχρι η ώρα να φτάσει 11 παρα 5. 12 συγγνώμη παρα 5, 12 παρα 5. Παρακαλώ ωστόσο όλοι να είστε εδώ κατά τις 12 παρα ώστε να είναι και αξιοπρεπή η υποδοχή που θα επιφυλάξουμε στον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.